Ο Κρίτσκο είναι πολύ γνωστός μποξέρ από την Ουκρανία, αλλά δεν υπάρχει μόνο αυτός. Ε, ευχαριστούμε κύριο κύριος Κίλαμ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε.